Συζητήσει μας. Τώρα έχω στην ημερήσια ένταξη τη λαοκρατική δημοκρατία του Κονγκό με τον κύριο Σεβαστιαν Η κατάσταση στην δημοκρατία του Κονγκό είναι σοβαρότατη. Αυτά τα οποία κάνει ο Καμπιλά για να παραμείνει στην εξουσία, ενώ το εμποδίζει αυτό το σύνταγμα της χώρας του δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταστέλλονται οι διαμαρτυρίες αυτές και προκαλούν πάρα πολλά θύματα ακόμα και θανάτους. Αυτό οδηγεί στην πτωχοποίηση, την τεράστια φτώχεια που χτυπά το σύνολο του πληθυσμού της χώρας και οδηγεί επίσης και σε αυτόν τον εσωτερικό πόλεμο χαμηλής έντασης ανάμεσα στους πληθυσμούς του Βορρά και του Νότου και που χτυπά κυρίως τις γυναίκες η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων ε, υπογράφει την πρόταση αυτή για να απαιτήσει από τον Καμπυλά να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και να κατανοήσει ότι δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία ενάντια στο Σύνταγμα και ενάντια στην βούληση του λαού θα πρέπει όμως να υπάρξει και μία αναφορά στο θέμα της εμπορίας των ορικτών από ζώνες σειράξεων και συγκρούσεων. Δεν υπάρχει ένα εμπόριο αίματος θα έλεγα για κάποια ορυκτά, για κάποιες ορυκτές πρώτες και θα πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Ο κύριος Ντεμασμάκερ. Έχουμε φτάσει σε μία περίοδο κέρια για την ε, λαϊκή δημοκρατία του Κόγκο οργανώσει των πολιτών, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ακόμη και εταίροι του Καμπυλά ζητούν αλλαγές ε, και αντικατάστασή του στην εξουσία. Αλλά εκείνο επιμένει να παραμένει στην εξουσία, παρότι είναι αντίθετο αυτό με το Σύνταγμα. Η κατάσταση πολιτική επιδεινώνεται, είναι ε, η ηλικιώδη ταχύτητα με την οποία επιδεινώνεται η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν έχει κανεί το δικαίωμα να μιλάει. Δημοσιογράφοι, οργανώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, φυλακίζονται, δολοφονούνται, διώκονται με κάθε τρόπο. Ακόμα και νέα παιδιά ε, το Φρέγκο Μάλι θα σας αναφέρω παραδείγματα που βρίσκεται στη φυλακή πάνω από ένα χρόνο περιμένοντας την δικαστή Πρέπει λοιπόν να δεδεμαστήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ουσιαστικό ρόλο για να ξεκινήσει ένας ανοιχτός διάλογος ε, για να προχωρήσει το Κονγκό, ε, να γίνει ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος δημοκρατικό, που το οποίο θα συμβάλλει και στην ειρήνη που τόσο περιμένουν οι Κονγκολέζοι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοράου, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η δημοκρατία του Κόγκο αντιμετωπίζει μια τεράστια πολιτική κρίση που απειλεί τη δημοκρατία. Βλέπουμε ποια είναι η απόπειρα του Καμπιλά να παρατείνει την εντολή του μέσω της καθυστέρησης της εκλογικής διαδικασίας παραβιάζοντας το Σύνταγμα και παραβιάζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι μια χώρα εμβληματική της ανυπαρξίας συνοχής της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης είναι η πιο πλούσια πάντα χώρα σε επίπεδο πρώτων υλών. Βλέπουμε τις εμπορικές συναλλαγές που έχουμε με τη χώρα αυτή και θα πρέπει εμείς να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του σεβασμού των συνταγματικών ρυθμίσεων και αν θα υπάρξουν πραγματικά ελεύθερες εκλογές χωρίς παράνομη παράταση ε, της θητείας του Καμπυλά και θα πρέπει να απελευθερωθεί και ο υπεύθυνο γκοή τη αντιπολίτευσης για να προχωρήσει σε θεραπεία διότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο κύριος, η κυρία Γκάμπριελ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι που έχουμε σήμερα αυτό το κατεπήγον ψήφισμα που θα συζητήσουμε την προεκλογική διαδικα... Ε, κατάσταση στην λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Οι επόμενοι μήνε έχουν κρίσιμη σημασία και για το μέλλον τη ίδια τη χώρα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή των μεγάλων λιμνών. Ε, υπάρχουν βασικά στοιχεία λοιπόν που θέλω να τονίσω. Πρώτον, όσον αφορά τη διαδικασία την εκλογική, θέλουμε την ε, τήρηση των προποθέσεων που έχει διατυπώσει η Επιτροπή Παρατήρηση των Εκλογών του 2011 και αργότερα η επίσκεψη, ε, τα αποτελέσματα της επίσκεψης, οποίας είχα την τιμή να ηγηθώ. Χρονοδιάγραμμα για τις εκλογές, προϋπολογισμό για τις εκλογές, ε, δέσμευση για σεβασμό ε, αμελητή του συντάγματος προκειμένου να μην κυλήσει στη βία η χώρα. Δεύτερον, πρέπει να ανανεωθεί βεβαίω για λόγου ανθρωπιστικού η παρουσία τη UNESCO και η προστασία στου πολίτε η περιφερειακή διάσταση ευρωπαϊκή αλλά και η, και Αφρικανική Ένωση πρέπει να, να αναπτύξουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διαφυλαχθούν οι σχέσεις και να αποκλειστεί η αδίποτε περίπτωση κλιμάκωσης της βίας στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Γκέρεν. Ε, οι συνταγματικέ διατάξει ε, πρέπει να προστατεύουν ε, του πολίτε κράτου από τι αυθαιρεσίε των ηθινών και σπάει η εμπιστοσύνη όταν δεν τηρούνται αυτές οι διατάξεις. Και αυτό γίνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Αναβάλλονται εκλογές τάχα για να ε, τροποποιηθεί το Σύνταγμα. Ο στόχος είναι ο περχόμενος πρόεδρος να παραμείνει για τρίτη ε, θητεία. Αυτό ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε τελικά εδώ στην Ολομέλη για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Και ναι, πιστεύω ότι πρέπει. Γιατί, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ στενά παρακολουθεί τη μεταβατική διαδικασία για Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από την αρχή έχει ε, πιστεύω συνεισφέρει ε, στο να υπάρξουν απαραίτητε προϋποθέσεις για τις εκλογές που έγιναν. Στήριξε, προσπάθησε να στήριξει τη δημοκρατία, κάτι που ζητούν και οι Κογκολέζοι. Επομένω, το Κοινοβούλιο ε, συνεχώ πενθυμίζει στις αρχές της Δημοκρατία από τι δεσμεύσεις τις οποίες έχουν αναλάβει και πρέπει να τηρούν. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη η κυρία Σέντρα Ροντρίγκεθ. Ευχαριστώ πολύ το ψήφισμα. Νομίζω ότι είναι ασθενές και γι' αυτό θα πρέπει ε, να εμβαθύνουμε σε κάποιες ακόμη πτυχές που ε, έχουν να κάνουν με τις καταπατήσεις των δικαιωμάτων στο Κονγκό. Πιστεύω το κοινοβούλιο μας θα πρέπει να εγκρίνει μέτρα τα οποία θα θέσουν ένα τέρμα ε, στις ευθύνε των πολιεθνικών και στην χρηματοδότηση της ενόπλης σύραξης. Τον Απρίλιο του 2015 γενικός, συγγνώμη, ο Διευθυντής του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον έλεγε ότι το 2% των κερδών από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων ε, ουσιαστικά πηγαίνουν ε, στα χέρια των ένοπλων ε, αυτών ομάδων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν μέτρα για την αναθεωρήση και για την αποκλήση από συμβάσεις εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου δασικού και ορυκτού. Και τέλος πιστεύω θα πρέπει να μιλήσουμε ότι θα πρέπει να πάψει η ε, αρπαγή γεών από τις πολυεθνικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, πρόεδρος Αρενά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το Σύνταγμα του Κονγκό προβλέπει ότι πρέπει να γίνουν εκλογές μέσα στι προσεχείς 90 ημέρες, οπότε, οπότε και εκπνέει η εντολή του Πρόεδρου Καμπυλά. Ωστόσο, αυτό διατηρεί τη σιωπή του και φαίνεται ότι το σύστημα είναι διατεθειμένο να διατηρήσει την θέση του στην εξουσία. Κίνδυνο μεγάλο για τη δημοκρατία του Κόγκο. Υπάρχουν από το 2012 ιδιαίτερε πιέσει εναντί ασδήποτε φωνή αντίθεση στο καθεστώ. Ζητούμε λοιπόν με το ψήφισμα πρώτον το ταχύτερο δυνατό να εγκαθιδρυθούν οι όροι για τη διεξαγωγή ανώθευτων διαφανών και ελεύθερων εκλογών. Ε, η Αφρικανική Ένωση πρέπει να το ρόλο τη, δηλαδή να κάνει σεβαστό το Σύνταγμα και τις διαδικασίες, μια διαδικασία σαφή, στοχευμένη και καλούμε τα Ηνωμένα Έθνη να, να διατηρήσουν ενισχύ το, ε, την εντολή της Μενούσκο. Ευχαριστώ πολύ, Πρέντα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιμείνω στην ανάγκη διοργάνωσης ε, βουλευτικών και προεδρικών εκλογών πριν τα τέλη της χρονιάς στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αυτό προβλέπει το Σύνταγμα και πιστεύω ότι θα πρέπει αυτή τη γραμμή να ακολουθήσουμε. Απαρέγκλητα. Ο πρόεδρος ε, Καμπιλά έχει ε, να επιλέξει μεταξύ του σεβασμού του συντάγματος, άρα δύο θητείες το πολύ, και της ε, προσπάθειας να παραμείνει με κάθε τίμημα στην εξουσία. Εγώ ελπίζω να επιλέξει την πρώτη οδό, δηλαδή το σεβασμό του συντάγματος, διότι διαφορετικά φοβούμε ότι το σενάριο του Μπουρούντι και άλλων χωρών παρόμοιων θα επαναληφθεί αυτή, αυτός ο πειρασμός ε, ε, το δυνικές παραμονή στην εξουσία ξέρουμε που καταλήγει. Ευχαριστώ. Κυρία Κιέγγε, ένα λεπτό. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Οι προεδρικές εκλογές στη Δημοκρατία του Κονγκό είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι μια δημοκρατική πρόκληση. Η χώρα πρέπει να αποδείξει ότι σέβεται το Σύνταγμα και τις προβλέψεις του Συντάγματος που περιορίζουν σε δύο θητείες την Προεδρία. Θα πρέπει να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα εκλογικό με σεβασμό των αρχών του συντάγματος ζητώντας από ε, την κυβέρνηση να σεβαστεί την ελευθερία του τύπου είναι το ελάχιστο της δημοκρατίας. Ε, το τέλος λοιπόν ε, του καθεστώτος Καμπυλά είναι κάτι το απαραίτητο και θα επηρεάσει θετικά τη σταθερότητα της περιοχής ευρύτερα. Απαιτείται επίσης και η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων που σέβονται το Σύνταγμα της χώρας και ζητούμε από την, από την Οργάνωση για την Αφρικανική Ενότητα να επιβλέψει την δημοκρατική μετάβαση. Ο κύριος Νάρτ, μιλώντας για την δημοκρατία του Κονγκό, είναι κάτι το ηρωνικό γιατί αυτή η δημοκρατία δεν ανήκει στο λαό, ανήκει στις ένοπλες ομάδες και στην κλεοπλεπτοκρατία είναι, υπάρχει μια μικρή μειοψηφία των, της φυλής των Μακόγκο που ελέγχει τη χώρα εις βάρος της πλειοψηφίας. Είναι κάτι το οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα αυτή στην τελευταία θέση της ανάπτυξης στον κόσμο. Έχουμε δώσει τα τελευταία χρόνια 100 περίπου εκατομμύρια βοήθεια ε, ε, δυστυχώς όμως δεν έχει βοηθηθεί η κοινωνία των πολιτών. Η κλεπτοκρατία εξακολουθεί να σοβεί στην συγκεκριμένη χώρα. Τα άρθρα 8, 9 και 67 ε, της Συμφωνίας του Κοτονού θα πρέπει να εξαρτήσει την βοήθειά μας προς τη χώρα με το αν η χώρα είναι πράγματι δημοκρατική. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η ασταθής ε, δημοκρατική κατάσταση και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη λαϊκή δημοκρατία του Κόγκο ουσιαστικά μας κάνει ε, να αφιβάλλουμε κατά πολύ ε, για την δυνατότητα εξαγωγής δίκαιων εκλογών. Βλέπουμε η δυνάμεις της αστυνομίας και επιβολής της τάξης να διαλύουν με βίο τρόπο τις διαδηλώσεις και τις διαμαρτυρίες και ο πρόεδρος Καμπυλά κάνει ό,τι μπορεί για να καθυστερήσει τις εκλογές και να παραμείνει στην εξουσία. Ε, οι ε, πλητοπαραγωγικοί πόροι της χώρας ε, δεν αξιοποιούνται για την ευημερία του πληθυσμού αλλά δημιουργούν διαφθορά μια νέα ε, εκλογική εφορευτική επιτροπή με μέλη από την κοινωνία των πολιτών και από την αντιπολίτευση θα πρέπει να επιβλέπει τις εκλογές του Νοεμβρίου που θα πρέπει να διεξαχθούν οπωσδήποτε τον Νοέμβριο και να είναι δίκαιες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος είναι από το 2001 στην εξουσία, στη λαϊκή δημοκρατία του Κόγκο. Με πολύ κατασταλτικό καθεστώς, πιέσεις, βία, πρέπει να προστατευτεί το Σύνταγμα και να γίνουν εκλογές. Αν δεν συμβεί αυτό δεν μπορεί να θεωρείται μέλος της κοινωνίας των δημοκρατικών κρατών, η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Είναι πλούσια σε ορυκτό πλούτο η χώρα. Αλλά δυστυχώς οι πολίτες της είναι πολύ πτυχοί. Πρέπει επίσης να συνεχίσει οι προσπαθίες του και ο οργανισμός των Ηνωμένων στην περιοχή υπέρ της δημοκρατίας και της ειρήνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Ε, γίνεται όμως μεγάλη οχλαγωγή στην ε, αίθουσα. Δεν έχω χρόνο, λόγω και της φασαρίας που γίνεται, να ακούσω όλους τους ομιλητές. Πετήρ, θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την ανησυχία μου για την ε, πολύ σοβαρή αυτή κατάσταση στο Κονγκό. 7,5 εκατομμύρια στο Κονγκό φαίνεται ότι δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό ή στην ε, νοσοκομιακή περίθλιψη αυτή τη στιγμή και πολλά είναι τα παιδιά που δεν μπορούν να πάνε σχολείο λόγω ε, των ε, διαφόρων συγκρούσεων ε, και των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Τρία εκατομμύρια είναι εκτοπισθέντες και άλλο μισό εκατομμύριο έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε γειτονικέ χώρες επειδή εκδιώχθηκαν. Περιμένουμε να γίνουν οι προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο και ελπίζουμε να είναι το πρώτο βήμα προς τη δημοκρατική μετάβαση μετά από πολυετή εμφύλιο πόλεμο και πολλά χρόνια πολιτικής αστάθειας. Όλοι μαζί θα πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς στις δημοκρατικές αυτές διαδικασίες του Κόγκο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, κύριος Δενάν, έχει το λόγο. Πρόεδρε, νομίζω ότι ο πρόεδρος Καμπιλά πρέπει να ρίξει μια ματιά γύρω του. Δυστυχώς είναι και άλλα παραδείγματα κρατών στην Αφρική αιωνίων προέδρων που προσπαθούν να απαλλαγούν από τα συντάγματά τους. Ο Πλέσταν Πορέο, παραδείγματι, στην Πορκίνα Φάσο πρόσφατα αλλά επικράτησε η βούληση του λαού και άρχισε να λειτουργεί μια δημοκρατική διαδικασία. Τα πλούτη του Κονγκό, γιατί υπάρχουν όντω, είναι πλούσια όντω η χώρα, πρέπει να κατανέμονται με βάση ένα δημοκρατικό καθεστώ στον λαό που υποφέρει τόσο πολύ σήμερα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει εταίρο τη Αφρική γιατί έχουν κοινό μέλλον και πεπρωμένο αλλά πρέπει ταυτόχρονα και να επαγρυπνεί για το σεβασμό τη Δημοκρατία στην Αφρική. Ευχαριστώ Πρόεδρε η Πρόεδρος. Ευχαριστώ τον κύριο Ντονανού. Και έτσι ολοκληρώνει η συζήτηση με τον Επίτροπο Χαν που θα λάβει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ησυχία. Παρακαλώ, μη θορυβείτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι πολύ καλή η ευκαιρία συζήτησης της κατάστασης στα ανθρώπινα δικαιώματα στη Δημοκρατία του Κονγκό και αναμένει την αποδοχή του ψηφίσματος που ασχολείται με τις πολιτικές διαδικασίες, την πορεία προς τις εκλογές και την κατάσταση στον τομέα του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών. Η χώρα αυτή είναι μια τεράστια χώρα με τεράστιες προκλήσεις, όχι μόνο η φτώχεια, όχι μόνο η ασφάλεια, το θέμα της βίας εις βάρος των γυναικών. Μερικές φορές η χώρα αυτή μετατρέπεται οι περιοχές της τουλάχιστον σε πεδία μάχης και αντιμετωπίζει συνεχώς κρίσεις. Η εύθραυστη ειρήνη στην ανατολική πλευρά της χώρας ε, εξαρτάται από την μεγαλύτερη ειρηνευτική δύναμη. Το Μινούσκο έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ εύθραυστη ε, κατάσταση μετά από τις τελευταίες εκλογές του 2006 υπήρξε κάποια πρόοδος, η οικονομία αναπτύχθηκε, κάποιες ένοπλες ομάδες στην ανατολική πλευρά της χώρας ε, αφοπλίστηκαν, και υπήρξε μία μικρή θετική εξέλιξη σε επίπεδο οργάνωσης του κράτους. Τώρα βρίσκεται σε, θα έλεγα, κρίσιμη στιγμή. Το 2016 θα έπρεπε να είναι μια χρονιά εκλογών, αλλά θεωρεί αντιπολίτευση και φοβάται ότι οι προθεσμίες οι συνταγματικές δεν θα γίνουν σεβαστές. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι εκλογές και ο δημοκρατικός τους χαρακτήρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση θα πρέπει να συμφωνήσουν σε όλα τα πολιτικά θέματα. Θα πρέπει όμως από κοινού να βρουν ένα οδικό χάρτη που να οδηγήσει ε, στην ψηφοφορία. Η δημοκρατία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ε, δυστυχώς όμως ε, οι διαμαρτυρίες οι ειρηνικές αντιμετωπίστηκαν με βίαιη καταστολή και οι δημοκρατικές ελευθερίες απειλούνται από τις δυνάμεις ασφαλείας. Υπάρχουν συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δικαστική εξουσία έχει λειτουργήσει δυσανάλογα αυστηρά. Στις 8 Μαρτίου υπήρξε μια δήλωση στην Κινσάσα που υπενθύμησε στην κυβέρνηση την ανάγκη να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της. Η πρόκληση είναι τεράστια. Η οικονομία έχει θυγεί από ε, πτωτικές τάσεις στις τιμές των πρώτων υλών και η παροχή υπηρεσιών ε, δυστυχώς ε, χειροτερεύει στην χώρα. Πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει στην ασφάλεια, στην ανθρωπιστική βοήθεια και στην ανάπτυξη. Έχουμε μία μακροπρόθεσμη εταιρική σχέση και θα πρέπει να βοηθήσουμε όχι μόνο σε επίπεδο υλικό, όχι μόνο να στηρίξουμε τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τους υπόλοιπους Αφρικανούς εταίρους και τη διεθνή κοινότητα. Εμείς θέσαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα πρώτα και πιο σημαντικά. Έχουμε εργαστεί στενά και με τα Ηνωμένα Έθνη ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, στην ε, δημοκρατία του Κονγκό. Θέλουμε να μην υπάρχει πλέον ατιμορρησία και να τερματιστεί η σύγκρουση. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου και με τις αρχές της χώρας. Συμπερασματικά, Πρόεδρε, θεωρούμε ότι θα είναι δυνατόν η χώρα αυτά να προχωρήσει και να περάσει από την έκθραστη κατάσταση στο σεβασμό του συντάγματος στο κράτος δικαίου. Το μέλλον της δημοκρατίας του Κονγκό ανήκει κυρίως και απόλυτα στους πολίτες της. Θα πρέπει η φωνή τους να γίνει σεβαστή και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να το πετύχει. Το ψήφισμα λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έρχεται σε εύθετο χρόνο και θα βοηθήσει ε, ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ και για την ειδική προσοχή που δείξατε στην ομιλία μου. Πρόεδρος, όντως και ζητώ συγγνώμη εκ μέρους των συναδέλφων. Όντως επικρατεί ο στην ε, αίθουσα όταν φτάνουν κάποιες εκατοντάδες συνάδελφοι ταυτόχρονα για τις ψηφοφορίες. Αυτά συμβαίνουν, δεν μπορέσαμε να σας ακούσουμε με ηρεμία και ησυχία. Έχουμε λοιπόν λάβει τα, τα σχέδια ψηφίσματος, ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και όσο νουπό θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Ψηφοφορία λοιπόν.